Είναι πολύ σημαντικό δυστυχώ το γεγονό και χρειάζεται να ρίξει μια ματιά και σε τέτοια πράγματα η Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.